και είναι διαθέσιμο. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, δεν ισχύει αυτό, άρα εγκρίνεται, εγκρίνονται τα πρακτικά. Πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσια διάταξης. Ε, πρόκειται για τη δική μου δήλωση για τον προϋπολογισμό του 2013. Δραστηριότητες της Επιτροπής Συνδιαλλαγής. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Την περασμένη Τρίτη το 12 ε, έληξε η προθεσμία των 21 ημερών ε, για την ε, συνδιαλλαγή. Η αντιπροσωπεία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν μπόρεσαν να βρουν κοινή συνένεση σε κοινό κείμενο. Και έτσι η διαδικασία του προπολογισμού για το 2013 με βάση την, το σχέδιο πρότασης της Κομισιόν δεν κατέληξε σε συμφωνία έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την συνθήκη, τώρα η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει νέο σχέδιο προπολογισμού. Ήδη η Κομισιόν ανέφερε την Παρασκευή της τρέχουσας εβδομάδας, δηλαδή στις 23 Νοεμβρίου, θα καταθέσει τη νέα της πρόταση με την ελπίδα ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που είναι οι δύο ισότιμες ε, αρχές ε, που ασχολούνται με τον προπολογισμό να βρουν μια συμβαστική λύση η οποία θα ε, είναι η λύση για τον τακτικό προπολογισμό του 2013 που θα ξεκινήσει τον 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Να ξεκαθαρίσω ότι το Κοινοβούλιο φυσικά είναι, συνειδητοποιεί την ε, ευθύνη του για τον προπολογισμό και ζητά μία ε, συνένεση και με, ως προς την πρόταση της Κομισιόν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνένεση θα έχουμε ένα δεύτερο προπολογισμό. Αυτό είναι ένας από τους ε, τρόπους που μπορούμε να ακολουθήσουμε για τον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά δεν είναι ιδανική λύση. Έτσι λοιπόν Δεν θα λέγαμε όμως ότι θα είχαμε συνένεση με κάθε τίμημα. Τα τελευταία χρόνια είχαμε διασφαλίσεις από τα κράτη-μέλη, τις οποίες εμπιστευτήκαμε, ότι οι θέσεις του Συμβουλίου για τις ε, πληρωμές, που ήταν κάτω από την πρόταση της Κομισιόν, ότι οι θέσεις αυτές θα γινόταν αποδεκτές. Αυτό το κάναμε. Αναγνωρίζοντας ε, τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλά από τα κράτη-μέλη μας. Όλα τα θεσμικά οργανά ε, ήξεραν ότι η Ένωση με ε, τα επίπεδα που, ε, πληρωμών που είχε δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα και γι' αυτό το λόγο στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο όταν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις για το προϋπολογισμό του τελευταίου έτους, του προηγούμενου έτους είχε διακηρυχθεί πανηγυρικά ότι όλες οι πληρωμές που δεν θα μπορούσαν να ισοσκελιστούν με τους ε, ε θα μπορούσαν να προχωρήσουν χωρίς ε, μεγάλο πρόβλημα. Στην πανηγυρική δήλωση και τα δύο ε, και οι δύο αρχές του προϋπολογισμού, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, διασφάλισαν ότι θέλουν αυτά να τα κάνουν γρήγορα και χωρίς μεγάλα προβλήματα. Να σας διαβάσω αυτή την δήλωση και αναφέρω το αγγλικό κείμενο. Λαμβάνοντας υπόψη ε, τις συνεχές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης στα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν για μία μείωση του επίπεδου των πιστώσεων πληρωμών για το 2012 σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζητούν από την Επιτροπή να ζητήσει περαιτέρω πιστώσεις πληρωμών σε έναν διορθωτικό προϋπολογισμό εάν αυτές του 2012 δεν επαρκούν. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβουν θέση για οποιοδήποτε διορθωτικό, σχέδιο διορθωτικού προλογισμού όσο πιο γρήγορα γίνεται για να μην υπάρχουν κενά στις πιστώσεις πληρώμων. Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι μια δήλωση βουλευτών απλώς, είναι ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την θέση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η Κομισιόν ε, για το 2012 για τη συνοχή, τα κοινωνικά ταμεία, την ε, επιστήμη, τα προγράμματα Εράσμους έχει λογαριασμούς που δεν μπόρεσαν να ισοσχελιστούν 9 δις ευρώ. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά ε, την ανάγκη για περαιτέρω ε, πληρωμές για το 2012. Αυτό το αναφέραμε την 31η Οκτωβρίου, όχι με βάση εκτιμήσεις, αλλά με βάση νομικές ε, υποχρεώσεις που έπρεπε να πληρεί η Κομισιόν για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε σοβαρά για το προπολογισμό του 2013 πρέπει να κλείσει πρώτο σωστό ο προπολογισμό του 2012. Αν δεν διαπιστώσουμε ε, ε θα είναι, πόσοι θα είναι οι ανοιχτοί λογαριασμοί τον 31η Δεκεμβρίου του 2012 δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σοβαρά ποιον προϋπολογισμό χρειαζόμαστε για το 2013. Τα κράτη-μέλη Είπανε λοιπόν ότι μέχρι το τέλος της ε, διαδικασίας διαβούλευσης θα διασφαλίσουν ότι ε, θα έχουν μια δήλωση ε, ότι θα παραμείνουν στην δήλωσή τους του Νοεμβρίου του 2012 για τα 9 δις που λείπουν. Δεν μπορούμε να δώσουμε λοιπόν ε, την έγκρισή μας ε, με τον παραδοσιακό τρόπο. Όταν μιλάμε για νέα δις, ε, μπορούμε να προσφέρουμε 3, 4, 5 δις ως εναλλακτική. Αυτό το κάνανε τα κράτη-μέλη με αυτή τη βάση λοιπόν δεν μπόρεσε να βρεθεί κοινή λύση με το ε, Κοινοβούλιο γιατί αυτό που μας ζητούν τα κράτη-μέλη δεν είναι διαφορετικό από το να ψηφίσουμε έναν ελληματικό προϋπολογισμό. Το Κοινοβούλιο δεν είναι λοιπόν έτοιμο να ε, χειριστεί με έναν τόσο μη σοβαρό τρόπο ε, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και να περάσει αυτό που κάνουν τα κράτη-μέλη στο σπίτι τους στην Ευρώπη. Αν δεν βρούμε μια λύση για τον προπολογισμό του 2012 και υπάρχουν κάποιες, πολλές, ανοιχτοί λογαριασμοί που περάσουν μετακυλιστούν στο 2013, τότε το 2013 θα βρεθούμε ενώπιον δυσεπίλητων προβλημάτων. Κυρίες και κύριοι, αυτός, αυτή δεν είναι πλέον η τακτική διαδικασία προϋπολογισμού. Δεν πρόκειται για ε, μια σωστή δημοσιονομική ε, διαχείριση στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι ο προϋπολογισμός για το 2013 θα πρέπει να επαρκεί για να καλύψει όλες τις πιστώσεις πληρωμών για το επόμενο έτος. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που απομένουν από το 2012, όπως η κάλυψη των μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του τρέχοντος έτου. Πρέπει αυτά να τα συμπληρώσουμε με πλέον χρήματα. Πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτεραιότητες ανάπτυξη, ε, δυνατότητα ανταγωνισμού και απασχόληση θα παλέψει η πρόταση της Κομισιόν και για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων στην κατηγορία Α1 ε, μπορεί να κάνει βελτιώσεις. Ε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ήδη έχουμε διαπραγματευτεί επικοδομητικά και λογικά με το Συμβούλιο. Θέλουμε κι εμείς ένα προπολογισμό για το 2013. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, είμαστε ανοιχτοί και είμαστε και ελπίζουμε ότι με τη νέα πρόταση της Κομισιόν, έτσι όπως έχει γίνει ως τώρα η διαδικασία και στο Συμβούλιο, θα υπερισχύσει η άποψη ότι πρέπει κανείς να πληρώνει τους λογαριασμούς του. Ένα θετικό στοιχείο για το τέλος. Μπορούμε τουλάχιστον μέσα από την επιμονή του Κοινοβουλίου και εγώ προσωπικά έχω πολύ δουλέψει γι' αυτό και ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες, ειδικότερα τον συνάδελφο Λαμασούρ και τον ε, Λαβεμαβίαρ και την κυρία Παλτσάνη. Όλοι από κοινού παλέψαμε έτσι ώστε ε, να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 5 για το 2012 με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης για τους σεισμούς στην Ιταλία ε, πρέπει να ψηφιστεί άμεσα στο ύψος των 670 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι λοιπόν, ε, σήμερα το μεσημέρι δείξαμε ε, να δώσαμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης με τα κράτη-μέλη και με τους πολίτες τους. Ε, πριν από λίγα λεπτά υπέγραψα αυτόν τον διορθωτικό προπολογισμό του κ. Μαυρογιάννη, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να στείλουν το πραγματικό μήνυμα αλληλεγγύης σε αυτούς που επλήγησαν πιο πολύ στις κοινότητες της Εμίλια Ρωμάνα στην Ιταλία, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα χρήματα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι για τα υπόλοιπα θέματα τα δημοσιονομικά θα βρεθεί ε, μια τελική θετική λύση και ότι τον Δεκέμβριο στην Ολομέλεια θα μπορέσουμε να έχουμε τις επαρκείς αυξήσεις και στο ε, διορθωτικό προϋπολογισμό 6 για το 12 και θα έχουμε και έναν καλό προϋπολογισμό για το 2013. Στο τέλος κυρίες και κύριοι να πω ότι για μένα ως τώρα η διαδικασία αυτή του προϋπολογισμού ήταν ε, καινούργια γη, τουλάχιστον ως προς την υπό την αρμοδιότητά μου ως ε, πρόεδρος αυτού του σώματος. Έμαθα πολλά. Καταρχάς έμαθα πράγματα πολλά ε, για τη διαφορά μεταξύ των λέξεων Συμβούλιο και της πραγματικότητας των μελών. Το Συμβούλιο είναι ο κύριος Μαυρογιάννης, δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη, αλλά στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι έτοιμα να τηρήσουν τις δικές τους υποσχέσεις είναι κράτη-μέλη που είναι έτοιμα να μας ε, ρίξουν σε μια διαδικασία ελληματικού προϋπολογισμού. Αυτά δηλαδή που κάνουν πολύ συχνά στους δικούς τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Χαίρομαι που σπάνια ε, δεν έχουμε ε, παρόμοιες στάσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Τζοβάνι Λαβία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Μαυρογιάννη, κύριε και κύριε Επίτροπε, πράγματι την Τρίτη 13 έληξαν οι 21 ημέρες για την περίοδο συνδιαλλαγής, δηλαδή καταληκτική ημερομηνία από όπου μετά ε, βλέπουμε ότι δεν επήλθε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής για τον ε, προϋπολογισμό. Από την αρχή λοιπόν κατέστη σαφές και εμείς το έχουμε υπογραμμίσει ευθύ εξ αρχής και στις επίσημες αλλά και στις άτυπες συναντήσεις μας ότι δεν είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός του 2013 να αντιμετωπιστεί χωρίς να έχουν καθαριστεί οι λογαριασμοί για το 2012. Και επομένως θα πρέπει να εξετάσουμε εντελεχέστατα όλα τα προβλήματα που τίθενται με το διορθωτικό προπολισμό υπαριθμών 5 που σήμερα το πρωί εγκρίναμε στο Κοινοβούλιο, όπως είπε μόλις πριν ο Πρόεδρός μας. Πάνω απ' όλα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα είναι ο διορθωτικός 6 και ο προπολισμός του 2013. Ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη όπως προτάθηκε τη μεταφορά νέων από προηγούμενες δηλαδή περιόδους. Και έτσι ενδέχεται να έχουμε το πρόβλημα να καταφύγουμε στα δεκατημόρια. Εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε ε, σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, έχουμε και δικές μας προτεραιότητες που θέλουμε να απορασπίσουμε. Σε ό,τι αφορά στις πληρωμέ, για παράδειγμα, ζητούμε να υπάρχει ένα επαρκές επίπεδο πληρωμών για να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα τακτικά μας καθήκοντα και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές της Ένωσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να επενδύσουμε υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πρόκειται για προτεραιότητες και του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο τις έχει επιλέξει και αυτό προτεραιότητες του και στην ανάγνωση του προπολογισμού 2013. Φυσικά και έχουμε επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και θα τι λάβουμε υπόψη και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να θυσιάσει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βωμό της λιτότητας. Και χωρίς καμιά εξαίρεση όπως ζητούν ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις. Ε, ωστόσο, έχω και κάποια αισιοδοξία βλέποντας και την εξαιρετική συνεργασία, το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και έτσι αισιοδοξώ ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά όμω τώρα την διαδικασία αυτή, επαναλαμβάνω, ε, συναποφασίζουμε με το Συμβούλιο. Ορίζεται λοιπόν ε, η συναπόφαση ε, και δυνάμει της συνθήκης. Θα την αξιοποιήσουμε αυτή την εξουσία υπέρ των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Γκάρτια Θάμπαλ Ρουμπιάλ. Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σε αυτή τη συζήτηση πρέπει ουσιαστικά να μιλούμε για τη συμφωνία που επετέφθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον προπολογισμό του 2013. Αυτό θα έπρεπε να είναι το αντικείμενο τη συζήτηση. Δυστυχώ δεν είναι γιατί δεν υπήρξε συμφωνία. Ούτε καν η συζήτηση δεν έχει ξεκινήσει. Αυτό που περιμένουμε ακόμη λοιπόν είναι να αποφασίσει το Συμβούλιο να πληρώσει τα τιμολόγια που εκκρεμούν για το 2012. Όπως είπε και ο πρόεδρος Σούλτς, όπως είπε και ο εισηγητής για τον προπολογισμό του 2013, ο κύριος Λαβία, στο Κοινοβούλιο έχουμε μια πάρα πολύ ξεκάθαρη και πολύ λογική θέση. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε για τον προσέχη προπολογισμό αν δεν έχουμε λύσει προηγουμένω τα προβλήματα της τρέχουσας χρονιάς. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Είναι τιμολόγια Τη τάξη των 9 δι ευρώ που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί και με τα οποία πραγματικά ε, λόγω ακριβώ αυτή τη κατάσταση, πλήττονται εκατομμύρια πολιτών. Κύριε Μαυρογιάννη, 500 εργαζόμενοι από τη χώρα μου δεν μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση. Το ίδιο συμβαίνει και με 512 ιταλού εργαζόμενου. Ε, με 1.050 στην Αυστρία, 1.000 στην Φιλανδία, 1.900 στη Ρουμανία, 303 στη Δανία. Δεν επηρεάζονται όμω μόνο αυτοί οι εργαζόμενοι και οι φοιτητέ, οι σπουδαστέ, ε, δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουν να πάρουν υποτροφία εράσμου. Οι ερευνητέ από, από πανεπιστήμια, από επιχειρήσει δεν γνωρίζουν θα... κατά πόσο θα πληρωθούν για την εργασία που έχουν παράσχει. Και γιατί όλα αυτά. Γιατί δεν δέχεται να πληρώσει το Συμβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό δεν καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο διαπραγματεύσει και γι' αυτό σήμερα περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τη θέση του Κοινοβουλίου και περιμένουμε η πρότασή τη ε, να ευθυγραμμιστεί με, τα δικά μας, με τις δικές μας ε, προσδοκίες. Ελπίζουμε ότι υπάρχει περιθώριο ώστε να δοθούν πόροι μεγαλύτεροι, περισσότεροι για διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, την έρευνα, την ανάπτυξη, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ή για τα προγράμματα εκπαίδευση και κινητικότητα ε, για την νεολαία μα. Αυτά θέλουμε να προωθήσουμε, το έχουμε πει και σε άλλε συζητήσει μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλε διαφορέ ό,τι αφορά τι προτεραιότητε και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια ταχεία ικανοποιητική συμφωνία. Εκεί που κολλάει όμως το πρόβλημα πιο πολύ είναι το επίπεδο των πληρωμών. Αν δεν ε, έχουμε παράλυση προγραμμάτων, ανησυχία των σπουδαστών ε, για τι υποτροφίε του. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να μην αναθεωρήσει επιταχύρω τις προτάσεις της. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και για το 2013. Δύο χρόνια υποσχέσεων και μη τηρηθισών ε, υποχρεώσεων. Δεν μπορούμε να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση εάν δεν ε, δεσμευτεί το Συμβούλιο να ε, τα καταθέσει τα χρήματα. Το κάναμε μια φορά αυτό το λάθος, δεν θα το ξανακάνουμε το Συμβούλιο δεν τηρεί τι υποχρεώσει του. Και εδώ οφείλονται και τα προβλήματα. Κύριε Μαυρογιάννη, ελπίζω να καταφέρετε να καταλήξετε σε μια συμφωνία, γιατί αυτό είναι στα χέρια του Συμβουλίου πλέον. Thank Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μούλτερ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αποχώρησε ο πρόεδρος Σούλτσε, αλλά πιστεύω ότι εξέφρασε ορθότατα στα εισαγωγικά του σχόλια τα πεπραγμένα. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο γίνονται παραχωρήσεις από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι είναι υπερβολικές οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου, ότι έχει αλλάξει άρδινη συγκυρία και όλοι θα αντιλαμβάνονται ότι πλέον δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τα προσυμφωνηθέντα μέτρα. Όμως, όταν προσυπογράφετε μία σύμβαση και ω εκ τούτου λαμβάνετε μία υποχρέωση, δεν μπορείτε να ξαφνιάζεστε όταν αρχίζουν να έρχονται λογαριασμοί ή η η Έτσι είναι τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να υπερβούμε το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται ο πληθωρισμός. Πολύ φοβούμε ότι λόγω των προηγουμένων υποχρεώσεών μας θα πρέπει να κάνουμε τις πληρωμές. Το θέμα είναι αν είναι ορθές οι ε, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν πολλές σχετικές παρανοήσεις. Εάν βασιστούμε στα στοιχεία που καταθέτουν τα ίδια τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε δεν θα πρέπει να αναμένουμε 6 ή 7% αύξηση στον προϋπολογισμό, αλλά θα πρέπει να αναμένουμε τη διπλάσια αύξηση τώρα. Θα χρειαστεί στα κράτη-μέλη ένα είδος ε, επίσημου κρατικού οργανισμού που θα επαληθεύει τα στοιχεία που ε, καταθέτουν τα κράτη-μέλη. Πρόεδρε, έχω δύο λεπτά στη διάθεσή μου και όχι ένα. Συνεχίζω. Θα πρέπει λοιπόν να επαληθεύσουμε αν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις της Επιτροπής ε, είναι σωστές. Ε, εν τη αυτή περιπτώση δεν θα έπρεπε να δυσκολευόμαστε κάθε χρόνο για να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό. Ο μόνος τρόπος είναι η περικοπή των πιστώσεων. Σας ευχαριστούμε. Ένα λεπτό είχα τελικά. Ο κύριος Άσουαρθ, πρόεδρε. Η αποτυχία της συνδιαλλαγής, ε, κατά τη γνώμη μου, είναι λυπηρή η ανταπόκριση του τύπου ισοδυναμεί με ένα πάρα πολύ αρνητικό μήνυμα προ την κοινή γνώμη. Αυτό είναι ένα από του λόγου Δίνουν την εντύπωση ότι δεν συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν δεν λάβει περισσότερα κονδύλια. Ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, πρωτού αποχωρήσει από την αίθουσα τη Ολομέλεια, εξέθεσε με σαφήνεια την κατάσταση. Ε, είναι μια τεχνική εμπλοκή. Πρόκειται για 9 δις ευρώ, είναι το ποσό που αναφέρεται στο διορθωτικό ε, σχέδιο προϋπολογισμού υπαριθμών 6. Όπως είπε και ο κύριος Μούλτερ όμως, ε, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από το παρελθόν. Χρειαζόμαστε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερο έλεγχο σε σχέση με την εκτίμηση του κόστους και των δαπανών από πλευρά των κρατών μέλων. Στο μεταξύ, θέλουμε πάγωμα του προϋπολογισμού στα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2010 δεν μπορούμε να αναμένουμε αν είμαστε εχέφρονες, μία μεγάλη υποχρέωση που συνιστά υπέρβαση 20 δισεκατομμυρίων ε, για το νέο πολιετές ε, πλαίσιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να επιληθεί από το Συμβούλιο και πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να επιδιώξει μια δέσμευση από πλευρά του Συμβουλίου με στόχο την ε, πρόορη περάτωση της διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ανδρέα, η συνδιαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2013 απέτυχε στη Γέννα ήδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επιπροσθέτω 9 δι για να καλύψει τις αιτήσει πληρωμές του 2012. Εγώ χαρακτηρίζομαι από σκεπτικισμό για αυτά τα επιπρόσθετα κονδύλια. Ε, εν καιρό κρίση ε, δεν αντέχουν τη συγχρηματοδότηση τα κράτη-μέλη. Θυμηθείτε ότι το Φεβρουάριο του 2012, μετά το κλείσιμο και την εκαθάριση των λογαριασμών του 2011, ο Επίτροπο για το Προπολογισμό Επίτροπο μα είπε ότι έχουμε μία έλλειψη 9 δισεκατομμυρίων. Δύο μήνε μετά, τον Απρίλιο, μα είπε ότι έχουμε πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίου. Και στη συνδιαλλαγή αλλαγή. Την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Λεβαντόσχη για το 2012 μας μίλησε για ανάγκη περικοπής των πληρωμών κατά 1,5 δισεκατομμύριο. Ε, λοιπόν, ποια, ποιο πόσο πρέπει να πιστέψουμε κι εμείς. Ε, νομίζω ότι πλήττεται η αξιοπιστία μας ε, στα, στις διαπραγματεύσεις, κυρίως η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πρέπει να χορηγήσουμε επιπλέον κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι ότου να προσκομίσει αξιόπιστα στοιχεία. Το επαναλαμβάνω ε, εδώ και χρόνια αυτό το επιχείρημα. Σας ευχαριστούμε κύριος Μπουτικόφερ. Δέχεστε την μπλε κάρτα παρακαλώ. Σας δίνω το λόγο αξιότιμοι συνάδελφοι ρωτούν πώς ε, μέσα σε μια επιχειρηματική διαδικασία ένας ε, οφειλέτης ε, που του ζητάνε να πληρώσει τις οφειλές του, αυτός λέει ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτό, να το αντέξει. Δηλαδή, Ευχαριστώ. Το, ε, το μόνο, η μόνη συμβαστική λύση που δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι το ποσό του περασμένου Δεκεμβρίου για τον προπολογισμό του 2012. Το Συμβούλιο είπε ότι θα διοχετεύσει, αν συντρέξει η ανάγκη, περισσότερα κονδύλια μέσα στον προπολογισμό για απρόβλεπτε περιπτώσει, όπω παραδείγματο χάρη πλημμύρε στην Ιταλία. Όμω, το να βρει κανεί τα 9 δι που αντιστοιχούν περίπου στο 7% του συνολικού προϋπολογισμού για το 2012 είναι κάτι απαράδεκτο και καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει ε, καμία λογιστική, αξιόπιστη λογιστική μέθοδος που να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γκαρίγκα θέλει να παρέμει, δέχεστε την ερώτησή του. Κύριε Αντρέασεν, τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τα κράτη-μέλη και τα οποία έχουν δοθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρείται ότι είναι αρκετή απόδειξη ε, αξιοπιστίας ή όχι. Ούτε και αυτά. Ε, I believe. Κύριε Γκαριγκά, έχουμε τεκμήρια ότι παραστατικά μάλλον ε, που αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια. Ε, ε, δεν εμφανίζονται ξαφνικά νυχθημερών ανάγκες 9 δισεκατομμύριων ευρώ. Συγγνώμη κιόλα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαυρογιάννης τώρα από πλευράς του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, επίτροπε. Λυπούμαστε ιδιαίτερα που η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, η οποία συνήλθε μετά την τελευταία συνάντηση του Κοινοβουλίου τον Οκτώβρη, δεν μπόρεσε να ε, συμφωνήσει μέσα στις 21 ημέρες που προβλέπονται στη συνθήκη. Η Κυπριακή Προεδρία έκανε τα μέγιστα για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε. Δουλέψαμε σκληρά για να συμφιλειώσουμε θέσεις ακόμα και μέχρι τις τελευταίες ώρες. Όμως, στο τέλος έπρεπε να αποδεχθούμε ότι οι απόψεις των δύο θεσμικών οργάνων είχαν μεγάλη διάσταση και δεν μπορέσαμε να βρούμε τελικά μία συμφωνία. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι έδειξε Πώ είναι αρκετά ανοιχτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες της περίοδου συνδιαλλαγή. Μπόρεσε να κάνει κάποια πρόοδο και ειδικότερα ήταν έτοιμο να εγκρίνει ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, διαπραγμάτευσης, τον διορθωτικό απολογισμό 5 ε, για το 2012 σχετικά με την κινητοποίηση 670 εκατομμυρίων ευρώ για το, από το Ταμείο Αλληλεγγύης για την υποστήριξη της Ιταλίας χωρίς αλλαγές ως προς την πρόταση της Κομισιόν. Παρά τούτο, δεν μπορέσαμε να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζονταν τα θεσμικά όργανα για να μπορέσει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος στον προϋπολογισμό του 2013. Η εντολή της Επιτροπής Συνδιαλλαγής ήταν να βρει μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013. Παρόλα αυτά αποδείχθηκε αδύνατο να προχωρήσουμε και αυτό χωρίς πρώτα να έχει αντιμετωπιστεί το θέμα του ε, σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 6 με, ε, που ζητά 9 δις ευρώ σε επιπλέον πληρωμές ε, για φέτος. Σωστό ε, ήταν αυτό που είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, η κυρία Γκαρτρία Μπάλ, ότι είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη για τα προγράμματα Εράσμους και είναι επίγον το θέμα. Εμείς ε, είμαστε δεσμευμένοι ως προς το να τιμήσουμε τις υποχρεώσεις μας για πληρωμές. Όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα αν θέλουμε να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα που θα έχει τη συνένεση όλων. Αυτό ήταν και το χάσμα μεταξύ των θέσεών μας. Για μας υπάρχει αναπόφευκτος δεσμός μεταξύ του ε, σχεδίου διορθωτικού προπολογισμού για το 2012 και του προπολογισμού για το 2013 γιατί και οι δύο προπολογισμοί στοχεύουν στη συνέχιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων και τα δύο πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις συνεισφορέ των κρατών μελών. Φυσικά, του του λεχθέντος, να πω ξεκάθαρα ότι τιμούμε πλήρω και σεβόμαστε τα δικαιώματα και προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ουσία και τη φύση της δημοσιονομικής διαδικασίας, δηλαδή τη, τη συνομοθεσία, τη συναπόφαση, ακόμα και αν οι ορισμένε προποθέσει είναι υπο... ευνοϊκοί προ εσά. Ε, μας έχουν μείνει τώρα μόνο λίγες εβδομάδες μέχρι το τέλος του έτους. Περιμένουμε, όπως υπόθηκε, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού από την Κομισιόν, ε, το οποίο θα λάβει υπόψη το πρόοδο που έχουμε επιτύχει και θα συμφιλιώνει τις διάφορες θέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ξεκάθαρα θα προτιμούσαν να βρισκόμασταν σε διαφορετική κατάσταση από αυτή στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Όμως, έχω ακόμα ελπίδες ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε θετικό αποτέλεσμα στο σύντομο χρονικό διάστημα που, παραμένει, που απομένει. Η Κυπριακή ε, Προεδρία βασίζεται στη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επικοδομητικό διάλογο έτσι ώστε να έχουμε έναν προπολογισμό έτοιμο για να, από τις αρχές του επόμενου έτους. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, είμαι πεπισμένος ότι η συνολική αξιοπιστία μας θα διακυβευτεί εάν δεν ε, βρούμε συμφωνία δεν θα καταλάβει ο κόσμος γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για θέματα τόσο σοβαρά. Και είμαι όμως πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να περκεράσουμε τις δυσκολίες και να βρούμε ένα μια συμβαστική λύση. Εύχομαι ε, να υπάρχει επιτυχές αποτέλεσμα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. so Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χέντεγκάρτ, η Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι δυστυχώς ο κύριος Λεβαντόφσκι εκλήθη εσπεσμένο στι Βρυξέλλε για την προετοιμασία των εργασιών για το πολιτέ πλαίσιο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαίτερα πολύ άσχολο σε αυτόν τον καιρό θα τον εκπροσωπήσω εγώ. Όμως πρώτα απ' όλα σε ό,τι είπε και ο πρόεδρος της αρχή του παρατήρηση να πω ότι και εμείς ε, χαιρετίζουμε την έγκριση του διορθωτικού προπολισμού παριθμών 5 που θα έχει ως συνέπεια να δοθεί υποστήριξη ε, στους πληγέντες ε, στην περιοχή την Εμίλια Ρωμάνη. Και είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί με κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει βέβαια τη λύπη της για το ότι δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία στη περίοδο συνδιαλλαγής για τον περιπλησμό του 2013. Είμαστε όμως ε, πεπισμένοι ότι εξακολουθούμε να έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε λύση μέχρι τα τέλη του τρέχοντος και τις επόμενες ημέρες η Επιτροπή θα υποβάλει ένα νέο σχέδιο προπολογισμού όπως προβλέπεται από το άρθρο 314 της Συνθήκης. Υπάρχουν βέβαια διαφορές μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής όμως σημείωσε ήδη πρόοδο, εντόπισε δηλαδή θετικά στοιχεία συμβιβασμού για τον προπολογισμό του 2013. Η Επιτροπή λαμβάνει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία υπόψη και θα τα λέω υπόψη και κατά την προετοιμασία του νέου σχεδίου προπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ω Επιτροπή να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τον προπολογισμό του 2013 πριν τα τέλη του τρέχοντος και να μην προσφύγουμε τελικά στα 12 Το επίπεδο των πληρωμών πραγματικά είναι ένα εκρεμές ακόμη ζήτημα, πάρα πολύ σημαντικό. Στη διάρκεια της συνδιαλλαγής ε, ένα σκόπελος ήταν ε, οι ελλείψεις πιστώσεων πληρωμών στον προπολογισμό και οι πρόσθετες ε, πιστός πληρωμών που ζητήθηκαν για το 2013. Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τα μέτρα στα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, είναι καθήκον τη Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τι νομικέ τη υποχρεώσει ε, λόγω των δεσμεύσεων που ανέλαβε και στο πλαίσιο του τρέχοντος και των προηγούμενων προπολογισμών. Ο έκτο διορθωτικό προπολογισμό είναι επιτάπητο και υπάρχει γενική αποδοχή του ότι πρέπει τα τιμολόγια να πληρωθούν. Μια πω στην κυρία Αντρέασεν ότι δεν μιλάμε, μιλάμε για πραγματικά τιμολόγια, δεν μιλάμε για εκτιμήσει. Μιλάμε για πραγματικέ αναληφθήσει υποχρεώσει και είναι θέμα αξιοπιστία για το τι κάνουμε εδώ. Μια εύλογη λύση για να αντιμετωπίσουμε τι ε, ανάγκε πληρωμών για το 2013 είναι κάτι που πρέπει να ε, κάνουμε τώρα για να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μα. Ιδίω απέναντι σε εθνικέ και περιφερειακέ αρχέ που στον τομέα τη συνοχή και τη ανάπτυξη πέθρου έχουν ήδη ε, αναλάβει τι υποχρεώσει του. Επίση, να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στου στους φοιτητές, σπουδαστές περιμένουν τι υποτροφίε του, είτε από το ερευνητικό πλαίσιο, είτε από το Εράσμου. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα ρεαλιστικό επίπεδο πιστώσεων πληρωμών για να προωθήσουμε μέτρα ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασία. Είναι κοινή προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα αυτό. Πανέρχομαι στον περιπλησμό του 2013 και στο τι μελγενέστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει πάνω το δυνατό για να υποβάλει ένα νέο σχέδιο προπολογισμού που θα μπορέσει να αποτελέσει μια σταθερή βάση, γερή βάση εργασία για Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και ω διαμεσολαβητής Ειλικρινή θα προσπαθήσει να βοηθήσει ώστε να εγκριθεί ο προπολογισμό του 2013. Ήδη Αντιμετωπίσαμε το 2010 μια ανάλογη κατάσταση όταν είχαμε τον πρώτο προπολογισμό σύμφωνα με τη νέα συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας. Απέτυχε η Επιτροπή Συνδιαλλαγής, αλλά μετά όλα τα θεσμικά όργανα εργάστηκαν επικοδομητικά, εντατικά. Κατάφεραν λοιπόν να εγκρίνουν τελικά τον προπολογισμό του 2011 σε αυτό το χρόνο. Για να ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω απλά μόνο κάποιες από τις επιπτώσεις που θα έχει το να μην επιτύχουμε ε, δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτές τις επιπτώσει. Θα σας πω με μερικά παραδείγματα τι θα γίνει. Σημαντικά προγράμματα και δράσεις θα μπορέσουν ή θα καθυστερήσει η εφαρμογή τους ε, και αυτό θα επηρεάσει άμεσα τους δικαιούχους. Αυτό μεταξύ άλλων θα συμπεριλάμβανε καθυστερήσεις πληρωμών για τις ε, δαπάνες και τι άμεσες ενισχύσεις για τη γεωργία. 70-75% αυτών ε, πρέπει να καταβληθεί ε, του χρόνου Γενάρη και Φλεβάρη. Δεν θα μπορούν επίση τα ειδικά μέσα να κοιτοποιηθούν όπω ε, το Ταμείο Λεγγύη, το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση ή το αποθεματικό για κατεπίδουσα βοήθεια για περίπτωση έκτακτη ανάγκη. Ή ρυθμιστικοί οργανισμοί επίση που αυτή τη στιγμή καθίσταται επιχειρησιακοί και αυτοί θα αντιμετωπίσουν προβλήματα για να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο του. Όπω. Ε, ο οργανισμός ε, για τα συστήματα πληροφορικής ε, στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων που θα γίνει επιχειρησιακός στις επόμενες ημέρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο και η Κυπριακή Προεδρία γνωρίζω ότι αντιλαμβάνονται τους κινδύνους αυτούς και είναι διατεθειμένα και τα δύο όργανα να συνεργαστούν εντατικά τις επόμενες εβδομάδες ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος για μια καλή συμφωνία εκφράζω τι ειλικρινεί ελπίδε τη Επιτροπή για εξέβριση λύση. Χάρη στι κοινέ μα προσπάθειε νομίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε έναν συμφωνηθέντα προεπιλογισμό το 2013 για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκε οικονομική ανάπτυξη και να δείξουμε την ικανότητα τη Ένωση να αντιδρά. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε σε αυτού του δύσκολου καιρού στου πολίτε τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασούρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Πρόεδρε το, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Για τον προπολογισμό κατέδειξε ρεαλισμό και στις ευθύνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο συναπτά έτη η ενισχυμένη πλειοψηφία, ευρεία μάλλον πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχτηκε το επίπεδο πληρωμών που είχε εγκρίνει το Συμβούλιο Υπουργών χωρίς να προσθέσει ένα ευρώ. Στι ψηφοφορίε μερίμνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να προαγάγει τι πολιτικέ προτεραιότητέ του που ταυτίζονται με αυτέ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή Θεματολόγιο 2020 και το Σύμφωνο Ανάπτυξη Εσχάτω. Αυτή η αίσθηση ευθύνη σήμερα μα οδηγεί, όπω ακριβώ έκανε και ο Πρόεδρο Σούλτ, να πούμε ότι ο προπολογισμό το 2013 δεν μπορεί να συζητηθεί εάν δεν ασχοληθούμε με τι καθυστερούμενε οφειλέ του 2012. Κανένα από του 27 υπουργού ναι, δεν αμφισβητεί το ποσό των καθυστερούμενων οφειλών. 9 δι. Κάποιοι όμω δεν θέλουν να καταβάλουν την πληρωμή. Δεν θέλουν να εκταμιεύσουν τι πληρωμέ ε, για πλήρω περατοθέντα προγράμματα το 2012. Αυτή η συμπεριφορά αντίκειται στο δημοσιονομικό κανονισμό, αντίκειται επίση στον προπολογισμό του 2010, όπω ψηφίστηκε, διότι έχουμε την πίστοση ανάληψη συγγνώμη, την ανάλυση υποχρεώσεων στην οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρο Σούλτσε, δηλαδή να ψηφίζεται διορθωτικό σε προπολογισμό του 2012. Αντίκειται επίση στι συνθήκε, διότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένο ο προπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί με ισοσκελισμένο τρόπο, όχι μόνο να ή Δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το έτο με ένα χρέο 9 δι. Προσθέτω ότι προ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η άρνηση ε, πληρωμή των τιμολογίων μα αφαιρεί η αδίποτε αξιοπιστία για του μελλοντικού προπολογισμού Ταυτόχρονα, ο προπολογισμό του 2013 υπενθυμίζει αυτού που το ξέχασαν σε κάποιες πρωτεύουσε ότι σε δημοσιονομικά θέματα είτε διαπραγματευόμαστε για ένα χρόνο είτε για εφτά, τίποτα δεν είναι εφικτό χωρί τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, και εμπιστευόμαστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαιρετώ την νέα Επίτροπο αρμόδια, λέει σαρκαστικά ο μιλητής ε, για ε, ε, τα θέματα προπολογισμού. ελπίζω να λάβετε υπόψη τι απόψει μα, να διευκολύνετε τη διαδικασία και ευχαριστώ την Κυπριακή Προεδρία που είναι ιδιαίτερα δραστήρια και αναλαμβάνει τι απαιτούμενε πρωτοβουλίε. Ευχαριστούμε, κύριο Βόγκαν τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήμουν με την ιδιότητα του εισηγητή στη διαδικασία συνδιαλλαγής ε, για το κεφάλαιο του Κοινοβουλίου και για τα υπόλοιπα ε, κεφάλαια. Δεν συζητήσαμε καν αυτά τα θέματα, διότι συζητήσει για το διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 5 και 6 απορρόφησαν όλο το χρόνο. Πάντως, χαιρόμαστε που επίσης έχουμε καταλήξει σε συμφωνία και είναι ένα ηθικό ζήτημα, δεν είναι μόνο δημοσιονομικό. Με ικανοποίησε λοιπόν η έκβαση των διαπραγματεύσεων Δυστυχώ για το διορθωτικό προπολογισμό 6 δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν πληρούμε τι νομικέ υποχρεώσει μα και αυτό που ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι το μέλλον κάποιων προγραμμάτων και ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο το ίδιο θα συμφωνήσει στο εσωτερικό του ε, γιατί αυτό είναι προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε. Σε σχέση με τους υπόλοιπους ε, τομείς ε, του προϋπολογισμού, ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτό που κάναμε είναι να διατηρήσουμε την αύξηση σε 1,9% για του χρόνου και χωρίς να έχουμε περικοπές σε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Αυτό το ποσοστό καλύπτει και το κόστος για την Κροατία, καθώς και αύξηση των μισθών κατά 1,7% για τον πληθωρισμό. Εμ και μόνο 0,6% περικοπή σε πραγματικού όρου αναγκαστήκαμε να δεχτούμε. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι λοιπόν. Σε άλλου τομεί υπάρχουν και άλλα εκκρεμή ζητήματα. Το συνολικό επίπεδο των αυξήσεων που θα χορηγηθούν σε άλλα θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο θέλει γενική, γενικό πάγωμα του προπολογισμού για όλα τα θεσμικά όργανα. Ε, αυτό είναι λάθο γιατί κάθε θεσμικό όργανο έχει διαφορετικέ ανάγκε και θα πρέπει να εξετάσουμε κάποιε περιπτώσει και να χορηγήσουμε και αύξηση ορισμένε περιπτώσει, η οποία όμω δεν θα υπερβαίνει, ξαναλέω, το 1,9%. Ένα άλλο εκρεμέ ζήτημα είναι η αύξηση των μισθών κατά 1,7%. Αυτή τη στιγμή θα αποφανθεί και το δικαστήριο για αυτό το θέμα. Ε, πιστεύω ότι είναι συνετό να περιοριστούμε στην αύξηση του 1,7% και να μπει η αύξηση στο αποθεματικό. Αυτό έχει ε, σημασία διότι ε, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να επιστρέψουμε στην κατάσταση του Ιουλίου του 2007. Ακόμη και σε αυτό το στάδιο απευθύνω θερμή έκκληση στο Συμβούλιο να κάνει την υποχώρηση και να δεχτεί την αύξηση του 1,7% μέσα στο αποθεματικό το τονίζω. Είναι το είναι το που έχουμε να κάνουμε. Ο κύριος Αλβάρο δεν είναι στη θέση του, ο κύριος Μορκάντη. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Τάνοκ. Έχει μπλε κάρτα. Δεχόμαστε την κάρτα. Να παρακαλώ. Κύριε Βόρν. Σα εκτιμώ ιδιαίτερα όπω γνωρίζετε. Κάθε μέρα παίρνουμε το ίδιο αυτοκίνητο για να έρθουμε στο Κοινοβούλιο. Αλλά πραγματικά πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση, ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχουν παγώματα μισθών και άνθρωποι απολύονται στο δημόσιο τομέα εξαιτία των περικοπών και τη λιτότητα κάποιοι ευρωκράτε, α πούμε, να ζητάνε 1,9% αύξηση στο μισθό τους, θα έπρεπε να υπάρχει πλήρω πάγωμα σε απόλυτους ε, ε, όρους ε, μέσα στα πλαίσια των περικοπών που υφιστάμεθα αυτή τη στιγμή. Κύριε Σμόρμ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν έκανα κάποιο σχόλιο για την αύξηση του 1,7%. Αυτό που είπα είναι ότι το ΔΕΚ μάλλον θα εγκρίνει αυτή την αύξηση και γι' αυτό θα πρέπει να πληρώσουμε αυτή την αύξηση του 1,7% είτε θέλουμε είτε όχι. Άρα υπό αυτές τις περιστάσεις είναι σόφρον για το Κοινοβούλιο να βάλει αυτά τα χρήματα στο απεθεματικό και για τα άλλα θεσμικά όργανα να κάνουν το ίδιο και καλό θα είναι να αποδεχθούμε αυτή τη θέση. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στον κύριο Μοργάντη. Κύριε Πρόεδρε, η αποτυχία της συνδιαλλαγής έδειξε όλα τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη, ε, τα οποία δεν μπορούν να συνεχίσουν πλέον. Αντί να στέλνουμε χρήματα στο λαό που έχει πληγεί από τους ε, σεισμούς, ε, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ντροπιαστικά επεισόδια της ευρωπαϊκής ιστορίας. Τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τις απαιτήσεις της Κομισιόν. Φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου λοιπόν για την Ευρώπη. Ε, ένα πράγμα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Όταν έχεις μια δέσμευση πρέπει να την τηρήσεις. Έχουμε όλα αυτά τα προγράμματα που ήδη έχουν θεσπιστεί, έχουν ήδη ξεκινήσει και το Εράσμου χρειάζεται χρήματα για να συνεχίσει. Για το μέλλον καλό θα είναι να είμαστε περισσότερο ρεαλιστές και να τα κάνουμε όλα αυτά και να αποφασίσουμε τι είναι πραγματικά προτεραιότητα. Θεωρώ όμως ότι σε κάποια περίπτωση πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί όσο η κατάσταση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανεί δεν πιστεύει σε αυτή, ε, πέρα από τα κράτη-μέλη που τη θέλουν, αλλά δεν θέλουν να πληρώνουν για αυτή πλέον. Ευχαριστούμε. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2013 απέτυχαν και αυτό είναι λυπηρό. Η διάσταση απόψεων ανάμεσα στα δύο θεσμικά όργανα ήταν υπερβολικά ευρύες ούτως ώστε τελικά να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Όμως έχουμε λιματικό προϋπολογισμό και έχουμε πρόβλημα με την καταβολή των πληρωμών του 2012 και άρα θα πρέπει να βρούμε μια λέση. Ουδάλλως θέτουμε εν κινδύνο για το 2013 την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποζημιώσεις προς τα κράτη-μέλη για τις ε, ήδη εγκεκριμένες πληρωμές πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Αυτό σημαίνει στην περίπτωση του έρασμου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα και άλλε πολιτικέ που ενδέχεται να πληγούν αν δεν ε, ψηφιστεί ο επιπρόσθετο διορθωτικό προπολογισμό, ανάπτυξη τη υπαίθρου, κοινωνικό ταμείο, ε, το ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7 για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο θεματοφύλακας των ε, δημοσιονομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν καταφέρουμε στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής ε, να αρχίσουμε να συζητάμε καν τον περιπλησμό του 2013 αφού δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις θεσμές που έχουμε αναλάβει για το 2012. Είναι ανάγκη λοιπόν να εγκριθεί ένα ακόμα διορθωτικό προεπολισμό ύψου 9 δι ευρώ. Αυτό είναι προ το συμφέρον των κρατών μελών. Διότι τα κονδύλια αυτά θα γυρίσουν πίσω στα κράτη-μέλη με τη μορφή επανεπένδυση στο πλαίσιο των δαπανών ε, του Ταμείου Συνοχή. Θα είναι πόροι οι οποίοι θα δοθούν ε, στους ε, ερευνητές και στους φορείς που χειρίζονται τις υποτροφίες του Εράσμους. Αν καταλήξουμε λοιπόν με το 12 θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε και για τον προϋπολογισμό του 2013. Όμως πρέπει να είναι σαφές το εξή. Αν δεν υπάρξει επιπλέον συνεισφορά από τα κράτη-μέλη θα τρωθεί η αξιοπιστία μας. Και μπορεί μετά η Κομισιόν να βάλει και νομικές κυρώσεις πιστεύω. Euroopan Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν προπολογισμό για να μπορέσει να φέρει οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και να βελτιώσει την ισότητα και να κάνει κάτι για την ανεργία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παλέψει για να γίνουν αλλαγές, ε, οποιασδήποτε αλλαγές στον προπολογισμό. Αυτό που πρέπει να γίνει στην Ένωση είναι να διασφαλιστεί ότι θα τελειώσουν όλες οι καταχρήσεις των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στο λαό. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ευθυνό, δεν είναι απλό. Αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Τα κράτη-μέλη θέλουν σκληρή πολιτική για τον προϋπολογισμό. Μιλάνε για την ευθύνη. Εμείς πρέπει πραγματικά να προσέχουμε ε, τα χρήματα που παίρνουμε από τους πολίτες, γιατί αλλιώς θα πρέπει να γίνουν περικοπές στο τέλος πρέπει τελικά να ανοικοδομήσουμε όλη αυτή την ε, δομή, να την χτίσουμε με σωστό τρόπο, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχουμε υποχρεωθεί να διεξαγάγουμε συγκεκριμένα προγράμματα, τα έχουμε εγκρίνει, τα έχουμε ελέγξει και τώρα πρέπει να τα πληρώσουμε πρέπει να πληρώσουμε οπωσδήποτε. Το θέμα είναι πότε. Αν δεν γίνει στο 2012, στις διαπραγματεύσεις του 2012 θα περάσει στο 2013 και αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και γι' αυτό έχουμε τα ανώτατα όρια τα οποία έχουν δοθεί ως βάση και το θέμα των 12 τιμωρίων που θα μας ε, αναγκάσουν να ε, δώσουμε αυτά τα χρήματα ε, με πλειοψηφία δύο τρίτων των, ε, του, του, Συμβουλίου και, και πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν η στιγμή να δείξουμε στον ευρωπαϊκό πληθυσμό ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με τον προϋπολογισμό μας. Ειδικότερα σε ποιες κρίσεις που έχουμε ελλείμματα χρειαζόμαστε εδώ να συμφωνήσουμε ειδικότερα για προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και επιτρέπουν την ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε η κυρία Χόλμαρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους ότι οι παλιοί λογαριασμοί πρέπει να ισοσκελιστούν και πρέπει να διασφαλίσουμε ώστε να μην γίνουν πιο ακριβοί μέσα από τους τόκους, έτσι ώστε να είμαστε αξιόπιστοι ε, απέναντι στους πολίτες μας. Σε αυτούς που υποσχεθήκαμε με ασφάλεια και τελικά δεν θα τους δώσουμε τα χρήματα. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διατυπωθεί αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2013 έχουμε το πρόβλημα ότι αυτά που θα εναπομείνουν τελικά θα αυξήσουν και αυτόν τον προϋπολογισμό. Οι υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους θα περάσουν σε αυτό και αυτό θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις ε, ε, οικονομικές. Καταλαβαίνω την κρίση, αλλά πραγματικά αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να το κάνουμε μέσα σε ένα πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, να συζητήσουμε τις υποχρεώσεις για αυτό, αλλά για το παρελθόν δεν μπορούμε να τα λύσουμε αυτά. Το σωστό πρέπει να γίνει. Χαίρομαι ε, λοιπόν ε, και ευχαριστώ που υπάρχουν τόσο εντατικέ διαπραγματεύσεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε. Εδώ τελειώνει το, κύριο, το Catch the Eye και περνάμε στην Επιτροπή με την κυρία Χέντεγκαρτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όπως είπαμε πρώτο, πριν από το τέλος αυτής της εβδομάδας θα καταθέσουμε νέα πρόταση επί τη βάση των απόψεων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι είναι κρίσιμος ο παράγοντας χρόνος και είμαστε της άποψης ότι εάν υπάρχει πολιτική βούληση, ακόμη είναι εφικτό να ψηφίσουμε τον προπολογισμό που χρειαζόμαστε για το 2013 και συνάγω από την σημερινή συζήτηση ότι όλοι συνειδητοποιούν ότι αυτό είναι το ελάχιστο. Περιμένουν οι πολίτε από εμά αυτή τη στιγμή. Το να μην μπορέσουμε να συμφωνήσουμε θα είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά τις επόμενες εβδομάδες και του επόμενου μήνες που υπολείπονται. Κύριε Μαυρογιάννη, παρακαλώ, από πλευρά του Συμβουλίου. Thank you very much, uh, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ενθαρρυντική ανταλλαγή απόψεων. Όλοι θα προτιμούσαμε να ήταν αίσια η έκβαση των διαπραγματεύσεων μετά το πέρας περίοδου συνδιαλλαγής. Παρόλα αυτά όλοι επιθυμούν να επανέλθουμε στις συζητήσεις και είμαστε όλοι προσιλωμένοι ούτως ώστε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 12. Όντως, με εδώ πέρα στις διαδικασίες συνδιαλλαγής, ε, σηματοδοτείται μια κοινή προσπάθεια και δέσμευση για να μην εγκαταλείψουμε τις προσπάθειές μας και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε συμφωνία. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να εκφράσω την ε, ειλικρινή εκτίμησή μου προς τον Πρόεδρο Λαμασούρο και όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, ε, το, επι, ε, το επικοδομητικό τους πνεύμα και να απευθύνω και χαιρετισμούς προς τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι και την κυρία Χέντεγκαρτ. Είναι ιδιαίτερα σε η συγκυρία και δυσχεραίνονται οι διαπραγματεύσεις ως εκ τούτου, άρα χρειάζεται να καταβάλουμε όλοι κοινέ προσπάθειες ούτως ώστε να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του 2013. Η Κυπριακή Προεδρία και εγώ προσωπικά θα ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καταλήξουμε σε έγκριση του προϋπολογισμού και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδραματίσει σωστά το ρόλο του διαμεσολαβητή, κυρίως απευθύνομαι στον Επίτροπο Λεβαντόσκη, σε σχέση με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού που τώρα καταρτίζει, ούτως ώστε να διευκολύνει τις μεταγενέστερες συζητήσεις μας. Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την προσοχή και την κατανόηση που δείχνετε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν και την Επίτροπο και τους συναδέλφους για αυτή τη συζήτηση. Περνάμε τώρα στις προφορικές ερωτήσεις σχετικά με τη διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Ντόχα.